περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για να είναι η πρόκληση ικανοποιητική για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Έληξη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα περνάμε στο επόμενο μας θέμα. Η σημερινή διάταξη τη διακυβέρνηση του διαδικτύου έκθεση του κυρίου Σώσα στον οποίο δίνω αμέσως και το λόγο. Τέσσερα λεπτά κύριε Βάγνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκταση που είχα την τιμή να συντάξω σε στενή συνεργασία με τους κύριους συζητητές θέλει να ορίσει το ίντερνετ ως ένα διεθνές δημόσιο αγαθό το οποίο θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε με στόχο το κοινό το διεθνές κοινό συμφέρον πρέπει να εμποδίζει τον έλεγχο από οποιαδήποτε οργανισμό ή ομάδα οργανισμών και κάθε προσπάθεια των κρατικών ή υπερκρατικών αρχών που θα έχουν στόχο να ελέγξουν τη ροή της πληροφορίας ε, του δικτύου. Βασική μέρημνα της έκθεσης ήταν η θέση που στην παγκόσμια διακυβέρνηση του ίντερνετ έχει ο Οργανισμός για την Ανάθεση Ονομάτων και Αριθμών, το ICANN. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό οργανισμό που υπόκειται στην νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογραμμίσαμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα του οργανισμού αυτού δεδομένου του λεπτού ρόλου που διαδραματίζει. Εμείς υποστηρίζουμε την διατηρήσή του γιατί γενικά ήταν θετικός, ε, θετική η δραστηριότητά του. Προτείνουμε ωστόσο μια μεταρρύθμιση που θα επιτρέπει μεγαλύτερη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στα διοικητικά όργανα του ΆΙΚΑΝ. Το ίντερνετ ωστόσο είναι πάνω απ' όλα ένα βασικό εργαλείο για την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και την εκμετάλλευση αυτών από μια πραγματικά δημοκρατική πολιτική κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν σοβαρέ ε, σοβαρές εγγυήσεις κατά νέων μορφών επαγρύπνησης, ελέγχου και λογοκρισίας από πλευράς των δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, τόσο ώστε η ελευθερία πρόσβαση στο ίντερνετ και η προστασία τη ιδιωτική ζωής να είναι πραγματικές και όχι φαινομενικές. Ζητούμε ιδιαίτερα από τις κυβερνήσεις να μην περιορίζουν την πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω παρεμπόδισης, ε, λογοκρισίας, φιλτραρίσματος ή άλλων μέτρων και να μην αναφέρουν σε ιδιωτικούς οργανισμούς τις δραστηριότητες αυτές. Οι περιορισμοί που κρίνονται αναγκαίοι Φερρυπίν για την προστασία των ανήλικων πρέπει να περιορίζονται στο αυστηρό αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία πρέπει να θεμελιώνονται στο δίκαιο και να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας όπως ε, αν το υλοποίησε, το παρουσιάζει και το ΔΕΚ και το ΕΔΑΔ. Η πρόσβαση στο ίντερνετ πρέπει να διευκολύνεται για όλους τους πολίτες με αποτελεσματικό τρόπο και κυρίως χωρίς διακρίσεις ε, με ειδική προσπάθεια σε ό,τι αφορά τα άτομα που ζουν στις αγροτικές περιοχές με βάση αυτά που προβλέπει άλλωστε και η ψηφιακή ατζέντα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Υπογραμμίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται ενιαία και ισχυρή φωνή της Ευρώπης στη διακυβέρνηση του ίντερνετ τόσο στο ICANN όσο και στα άλλα διεθνή βήματα. Ιδίως στο φόρουμ για την διακυβέρνηση του ίντερνετ διότι το μέσο αυτό είναι ένα βασικό εργαλείο διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνία των πολιτών και ιδιωτικού κλάδου. Η επόμενη σύνοδος του φόρμα αυτού θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βίλνιους. Η σημασία του ε, δεν πρέπει να αγνοηθεί, από ε, δεν αγνοήθηκε. Στην έκθεση υποστηρίξαμε ε, σαφώς και προτείναμε κάποιες αλλαγές στη λειτουργία του φόρουμ αυτού. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να υποσπιστούμε τις αρχές της Ένωσης όπως εκφράζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης, ιδίω τις σχέσεις μας με χώρες αξί, οι αξίες των οποίων μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές της Ευρώπης. Το ίντερνετ, συναδελφοί, είναι ο ωκεανός, το ανοιχτό πέλαγος που θα ενώνει κυβερνήσεις και ελευθερία. Τελειώνω ευχαριστώντας του συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου στην διατύπωση της έκθεση αυτή και τους υπαλλήλου τη επιτροπή που ε, με βοήθησαν, που μου προσέφεραν ανεκτήμητη βοήθεια. Ευχαριστώ που με προσέξατε τέτοια ώρα που είναι. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τώρα μία σειρά ομιλητών. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Βος. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η σημασία του ίντερνετ ε, και βεβαίως αυτό σχετίζεται με το αμέσως προηγούμενο θέμα αυξήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Ολόκληρα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν, έχουν βασιστεί στην αδιάλειπτη παροχή του ίντερνετ ε, και έχουμε φτάσει να έχουμε και εκπαίδευση αλλά και υποκατάστατο των ε, κοινωνικών επαφών, και άλλες μορφές ιδιωτικής επικοινωνίας, οπότε έχουμε μία υποδομή η οποία μοιάζει πράγματι με ένα δημόσιο αγαθό, οπότε θα πρέπει να έχουμε και κάποιον λόγο. Βεβαίως η ελευθερία του ίντερνετ σημαίνει και καταχρήσεις, αλλά είναι και μια αυταξία την οποία θα πρέπει να διατηρήσουμε και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε online αυτό το οποίο απαγορεύεται offline. Αλλά βεβαίως ε, αυτό δεν γίνεται μέσω της αυτορύθμισης όπως θα επιθυμούμε. Οπότε από τη μία μεριά υπάρχει ελευθερία και από την άλλη η ελευθερία και η ιδιωτική σφαίρα. Αυτοί οι στόχοι δεν είναι αντιφατική μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την περτέρω εξέλιξη και να έχουμε λόγο σε αυτήν. Ευχαριστώ η κυρία Ρόιτεβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα το ίντερνετ ελέγχονταν χωρίς να εμπλακούν οι κυβερνήσεις. Αυτό πλέον δεν είναι αποδεκτό. Η κυβερνοτρομοκρατία, η επιρροή χωρών όπως η Κίνα απαιτούν γρήγορα βήματα. Σήμερα λόγο έχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και μιλάμε για το ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υπόκεινται στον νόμο της Καλιφόρνιας. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι εσωτερικές δομές των διαχειριστικών αυτών οργάνων του διαδικτύου. Πιστεύω όμως πως η διακυβέρνηση του διαδικτύου από ένα σώμα του ΟΗΕ δεν είναι ευέλικτη αρκετά λύση. Χρειάζεται ένας αποτελεσματικός μηχανισμός έφεσης και διαιτησία, παραδείγματο χάρη σε οποιαδήποτε απόφαση. Επίση να αυξηθεί το επίπεδο δημοκρατική εκπροσώπηση μέσω οργανώσεων χρηστών και άλλων που αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Και όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη η Κομισιόν. Ε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η χρήση του διαδικτύου είναι απολύτως απαραίτητη και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις δεδομένου του ότι μέσω του διαδικτύου απολαμβάνουμε πολλές υπηρεσίες και αγαθά είναι πλέον ένα δημόσιο αγαθό παγκόσμιο στο οποίο θα πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της πρόσβασης ε, και βεβαίως ε, υποδομές ειδικά στις ε, περιοχές της υπαίθρου των αναπτυσσομένων χωρών έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την ψηφιακή ψαλίδα στην Ευρώπη και στις άλλες περιοχές του κόσμου, το ψηφιακό αυτοχάσμα. Βεβαίω θα πρέπει να προστατεύεται η υποδομή από κυβερνοεπιθέσεις οποιασδήποτε φύσης και νομίζω πως σχετικές αυτές προσπάθειες θα πρέπει να συσχετιστούν με τα άλλα μέτρα προστασίας και βέλτιστων πρακτικών που υιοθετεί η διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ. Ε, ogromnie dziękuję. Chciałem pogratulować e, sprawozdania. E, jedną e, Θέλω να την, ε, τον εισηγητή για το κείμενο του. Η ψηφιακή ε, ατζέντα θα επιτρέπει τα επόμενα χρόνια να μπορεί κάθε Ευρωπαίος πολίτης να έχει πρόσβαση στο ευρωζωνικό ίντερνετ. Το θέμα που εξετάζουμε είναι σημαντικό. Η συμμετοχή θα πρέπει να μετέχει, να περιλαμβάνεται σε μια εταιρική σχέση και η μεταρρυθμίση να επιτρέπει στην Ένωση να είναι πλήρως, ε, πλήρης εταίρος που θα επιτρέπει τη λειτουργία του εργαλείου αυτού. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελευθερία του μέσου της δομής αυτής και να προσπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, φερρυπίν την προστασία των ανηλίκων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το θέμα των ε, τυχερών παιχνιδιών στο ίντερνετ. Πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο για τα στοιχεία αυτά, προσπίζοντας βέβαια πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι κυβερνήσει των κρατών μελών σίγουρα θα θέλουν να ελέγξουν το μέσο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εταίρος των καθορισμό των κανόνων αυτών. Ευχαριστώ. Κύριος Πάσκα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ε, το ίντερνετ είναι πηγή πληροφοριών, απείρων πληροφοριών. Πρέπει να δούμε και την αξία τους, γιατί συχνά πρόκειται περί παραπληροφόρησης μαζί βεβαίως με το ίντερνετ φτάνουν στα δωμάτια των παιδιών μας η πορνογραφία, τα τυχερά παιχνίδια, τέτοια πράγματα. Οπότε όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν μαζί με το άνοιγμα της αγοράς του διαδικτύου. Πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες του ανοίγματο αυτής της αγοράς και να γνωρίζουμε το εάν οι οικογένειες μπορούν να προστατεύσουν εαυτούς από αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω πως αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη και αυτών που δίνουν την πρόσβαση. Κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε. Το Ευρωκοινόβουλιο μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε προς όλα τα φόρα και πολλά τα κονσόρτσια ώστε να τυποποιήσουν το ίντερνετ. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την υποδομή και να προστατευτούμε και από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο καθώς και να εξασφαλίσουμε και τα προσωπικά δεδομένα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει στη διεθνή συνεργασία προς αυτό τον ε, στόχο και να έχουμε καλύτερη συνείδηση των εγκλημάτων στην κυβερνοχώρο και να είναι σαφής οι ευθύνες για την κάθε πλευρά των συμμετεχόντων στον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντική ακόμη η ηλεκτρονική υπογραφή. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή υποδομή ώστε να έχουμε διασυνοριακή διαλειτουργικότητα και ασφάλεια. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι να ενισχύσουμε, την εμπιστοσύνη του χρήστη ώστε να χρησιμοποιεί υπηρεσίε και προϊόντα θα πρέπει να πιστοποιήσουμε τις ιστοσελίδες από την άποψη της ασφάλειας. Και τώρα η Επίτροπος Κρόες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το έντονο ενδιαφέρον του Ευρωκοινοβουλίου για, τον σημαντικό, για το σημαντικό θέμα της διακυβέρνησης του διαδικτύου έχει υποστηρίξει και ενισχύσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα. Η δημόσια πτυχή της διακυβέρνησης του διαδικτύου έχει γίνει πιο ορατή και πιο σημαντική πρόσφατα καθώς αναπτύσσεται το διαδικτύο και γίνονται αντιληπτά τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Βάγνερ και, καθώς και τους βουλευτές που σχολίασαν τα διάφορα θέματα δημόσιας πολιτικής που εμπεριέχονται στην έκθεση. Το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιό έχουν παρόμοιες ιδέες, κυρία Πρόεδρε. Θα θυμόσαστε όταν παρουσίασα την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη ότι πολλά από τα θέματα που τίθενται σε αυτή την έκθεση αντανακλώνται ήδη στις αρχικές ιδέες. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η ανάγκη να εξασφαλίσουμε τις ευρωπαϊκές ιδέες όπως ακριβώς τονίσατε και να περιέχονται στην σφαιρικότερη συζήτηση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται υπόψη στο διεθνή διάλογο για τη διαχείριση αυτού του παγκόσμιου πόρου. Θα έχουμε λοιπόν επαφές μέσα στο πλαίσιο της ΕΚΑΠ αργότερα αυτό το μήνα στις Βρυξέλλες. Επίσης αναφέρθηκε ότι ένα άλλο σημαντικό γεγονός φέτος θα είναι σίγουρα το, ε, το Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου στο Βίλνιους το Σεπτέμβριο και χαίρομαι πολύ που το Ευρωκοινοβούλιο έχει την πρόθεση να συμμετάσχει με πολλούς βουλευτές και φέτος. Αντιλαμβάνομαι ότι στην Προεδρία θα επιλέξετε τους συμμετέχοντες της, ε, στην αντιπροσωπεία αλλά ελπίζω ότι κυρία σόσα ο κύριος Σόσα Βάγνερ ε, θα έρθει και αυτός μια και έχει εργαστεί επί του θέματος τα τελευταία τέσσερα χρόνια πράγματα, πράγματι έχουν προωθηθεί οι ευρωπαϊκές αξίες χάρη στο έργο σας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριοι βουλευτές θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη για τη θαυμάσια συνεργασία μεταξύ των οργάνων μας και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχόλιο του κυρίου Σόζα Βάγκνερ. Ένα συναισθηματικό σημείο έχουμε όντως εμείς την ευθύνη να, προστα... να προστατεύσουμε τους ανήλικους από τις καταχρήσεις στο διαδίκτυο και πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να πετύχουμε και δεν είναι εύκολο αυτό όχι επειδή δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα αλλά αυτοί που συμμετέχουν στη δημιουργία του προβλήματος πραγματικά είναι άνθρωποι που αλλάζουν δρόμο και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα ανά πάσα στιγμή. Βεβαίω η προστασία, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εξασφαλίσουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλες δράσεις κλειδιά που είναι σκόπιμο να προωθηθούν και διασυνδέονται με αυτό το θέμα. Τα αναφέρατε άλλωστε. Συμφωνώ με όσους είπα ότι στο ΙΚΑΜ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Βεβαίως ε, υπάρχει και νέα πρόκληση καθώς το διαδίκτυο πολλά μας προσφέρει αλλά έχει και τα αρνητικά του. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αρνητικά αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε σίγουρα καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Μια τελευταία αναγγελία. Η συνεδρίαση διακόπτεται για αύριο, 15 Ιουνίου, στις 9.